Señorías, reanudamos la sesión. En primer lugar, he de hacer dos anuncios. El primero es que... Καλησπέρα σας. Ας αρχίσει η συνεδρίαση. Ε, ο κύριος Σιγνάτη παρετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 23 Απριλίου και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού μας ε, λαμβάνουμε γνώση της απουσίας του από την ημερομηνία αυτή και μετά και θα ενημερώσουμε και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Δεύτερη ανακοίνωση. Ε, στην συνάντηση του Απριλίου η Νομική Επιτροπή ενέκρινε την διαπίστευση των συναδέλφων Μπαουτίστα και Λίπινων. Και επίσης προτάθηκε με ομόφωνη γνώμη όλων την έγκριση της εντολής τους. Και αν δεν έχετε κάποια ένσταση θα θεωρήσω ότι η απόφαση αυτή έχει επικυρωθεί. Και τώρα, σύμφωνα με την μερισσία διάταξη, προχωρούμε στην ε, συζήτηση εκθέσεως Κρόλη που αφορά τη διάρκεια προστασία του δικαιώματος της πνευματικής με μένων συγγενικο δικαιωμάτων. Πρώτα πρώτα ο κύριος συζητής έχει το λόγο, ο κύριος Κρόλη για τέσσερα λεπτά. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ή στην αίθουσα και ο κύριο Μακρύβη στην αίθουσα και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που βρίσκονται μαζί μα. Αυτή η παρέκταση τη προστασία του δικαιώματο αποτελεί κάτι που όλοι το θέλαμε, Κυρίω διότι πάρα πολύ.